ανώνυμα να κυκλοφορούν τα δεδομένα και να τα προστατεύουμε. Επίσης μην ξεχνάμε ότι η υγεία αποτελεί ένα προνόμιο. Μια δεύτερη πρόκληση είναι ότι και οι γιατροί και οι ασθενεί πρέπει να είναι πιο υπεύθυνοι. Αυτή η διευκόλυνση, ψηφιοποίηση τη υγεία δεν πρέπει να μα κάνει να ξεχνάμε ότι κάθε τεχνολογική πρόοδο με τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει έναν ε, γιατρό ο οποίος διαθέτει όλα τα δεδομένα και μπορεί να εξυπηρετήσει τον ασθενή. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μιχαέλα Σόντροβα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίε και κύριοι, υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα γιατί πιστεύω ότι η ψηφιοποίηση βελτιώνει την περίθαλψη, βελτιώνει επίση την πρόσβαση στον τομέα τη υγεία, αλλά και την αποτελεσματικότητα του κλάδου. Και είναι μία από τι λύσει όσον αφορά την έλλειψη ιατρικού προσωπικού ε, που ε, πρόβλημα θα οξύνεται όσο γυράσκει ο πληθυσμός. Οι σύγχρονες ε, τεχνολογίες αντικαθιστούν την φυσική παρουσία των ιατρών, ιδιαίτερα στην εποχή μας, όπου ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού προτιμάει να απευθύνει τις υπηρεσίε υγείας μέσω ηλεκτρονικών τρόπων. Αλλά υπάρχουν και οι μεγαλύτεροι σελικοί άνθρωποι που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με αυτές τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες. Άρα λοιπόν η διευκόλυνση του ψηφικού μετασχηματισμού στην υγεία δεν θα, μας κάνει, δεν θα πρέπει να μας κάνει να λησμονούμε ε, την δυνατότητα προσβασιμότητας και την προσωπική σχέση μεταξύ ασθενών και γιατρών. Η... Ο κύριος Σουέλη. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα να πω ότι ε, με θλίψη μου διαπιστώνω ότι μιλάμε για το τομέα της υγείας και της περίθαλψης, ένας τομέας ο οποίος αναπόκειται στην αρμοδιότητα των χωρών μελών κατ' ουσία. Και δεν μπορεί να είναι αποδεκτό η υγεία των πολιτών και το προσδόκιμο ζωής να εξαρτώνται από το πού γεννιέται ένας πολίτης, από τον τόπο γέννησης. Επίσης δεν είναι αποδεκτό όσον αφορά την ποιότητα της ιατρικής περίθαλψης να υπάρχουν μεγάλες ε, διαφορές στην ποιότητα αυτών των παροχών. Ε, υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ Δυτικής ή Ανατολικής Ευρώπης. Για παράδειγμα, ε, η Ουγγαρία. Γι' αυτό είμαι υπέρ ενός ε, ελάχιστου προγράμματος παροχής ε, περίθαλψης. Θα πρέπει να εκπονηθούν προδιαγραφές, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ένα επίπεδο σώτας μεταξύ όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πάλμερ. Ευχαριστώ υποστήριξα αυτό το ψήφισμα. Δεν έχω αμφιβολία ότι η τεχνολογία οι ψηφιακές εξελίξεις, η καλύτερη χρήση των δεδομένων μπορούν να βοηθήσουν όλο τον τομέα της υγείας και της περίθαλψης σε εθνικό, σε ευρωπαϊκό και σε τοπικό επίπεδο. Όμως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με αυτό το θέμα, να εξασφαλίσουμε τα αυστηρότερα μέτρα διαφύλαξης και την καλύτερη προστασία κάποιων από αυτά τα δεδομένα, κυρίως τα ατομικά στοιχεία για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τον καθένα. Όταν αυτά ομαδοποιηθούν σε επίπεδο πληθυσμού, μπορούν να βοηθήσουν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών υγεία, νέων θεραπείων και ενίσχυση των συστημάτων υγεία. Θα πρέπει να είμαστε όμω ιδιαίτερη προσεκτικοί. Ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πώ θα σκεφτόμαστε τα δεδομένα, πώ θεωρούμε ότι τα δεδομένα μπορούν να γίνουν εμπορικό προϊόν. Πρέπει να υπάρχουν μέτρα διαφύλαξη και προστασία για αυτά τα δεδομένα. Ευχαριστώ. Τελευταίο. Ο κ. Πιλικέλα Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα. Οι υπηρεσίες ψηφιακής υγείας βελτιώνουν την περίθαψη κυρίως στην ύπεθρο της Ιρλανδίας. Κυρίως όταν αφορά την ψυχική υγεία, στην Ιρλανδία ο κόσμος πρέπει να περιμένει επί μεγάλο χρονικό διάστημα για να δει το γιατρό του. Να δει σύμβουλο, να δει ψυχολόγο, να δει τον ψυχίατρό του. Λογικό είναι να παρέχονται ηλεκτρονικές υπηρεσίες συμβουλών. Αλλά τα θέματα της ψυχικής υγείας δεν απαιτούν πάντα ένα ραντεβού που να βλέπει κανείς πρόσωπο με πρόσωπο το γιατρό του. Εξίσου αυτές οι υπηρεσίες εξαρτώνται από ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλή ταχύτητα που θα πρέπει να θέσουμε στην Ιρλανδία. Η Ιρλανδία κινείται, η Ιρλανδική κυβέρνηση, όσον αφορά την ευρυζωνική, κινείται με πολύ αργού ρυθμού. Χωρί ένα καλό σχέδιο, αυτέ οι ψηφιακέ ε, υπηρεσίες υγείας δεν θα διαθέσιμε στην Ιρλανδία όπως τα άλλα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Äh, Αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώσαμε αυτή τη διαδικασία επεξήγησης ψήφων και εδώ διακόπτεται η συνεδρίαση μέχρι τις 3 και εύχομαι στους παρόντες συναδέλφους καλή όρεξη. Mm -hmm. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπότιτλοι AUTHORWAVE

Πανί Good afternoon, colleagues. Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Αρχίζει η συνεδρίαση. Τα χτεσινά πρακτικά και τα κείμενα που εγκρίθηκαν είναι διαθέσιμα. Υπάρχουν σχόλια, οπότε εγκρίνονται τα πρακτικά. Πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη σήμερα είναι συζήτηση για τη συμβατότητα ανάμεσα στην ισχύουσα Συμφωνία Ελεύθερων Συνελεγών Ευρωπαϊκή Ένωση Μαρκοσούρ και την πρόταση τη Επιτροπή για μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Ενημερώνω του Ευρωβουλευτέ ότι δεν προβλέπεται διαδικασία κατσδιά σε αυτή τη συζήτηση και δεν θα δεχτούμε ούτε μπλε κάρτε. Αρχίζουμε λοιπόν με τον συντάκτη, τον κύριο Ζαντό. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο, κύριε Ζαντό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε κύριε Πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, για τους οικολόγους η Πράσινη Συμφωνία το να βρίσκεται στην καρδιά της ευρωπαϊκής ατζέντας καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και μια μεγάλη επιτυχία για τους επιστήμονες που εδώ και χρόνια κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Είναι μια μεγάλη επιτυχία επίσης για τους πολίτες που κινητοποιούνται, για τις επιχειρήσεις που αρχίζουν να δρούν. Αποτελεί βέβαια και επιτυχία για τους οικολόγους μετά τις τελευταίες εκλογές και αποτελεί και επιτυχία βέβαια για την παγκόσμια νεολαία που επίσης κινητοποιείται για αυτά τα θέματα και που ζητάει δράση από εμά. Αλλά πρόκειται και για μια τεράστια ευκαιρία. Ευκαιρία για την Ευρώπη να έχει στη διάθεσή τη ένα κοινό ορίζοντα, ένα κοινό σχέδιο, να βοηθήσει το κοινό υπέρ τη καινοτομία, της ε, ε, ε, κοινωνική, της δημοκρατικής, για την οικονομία μας, για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης στην επικράτειά μας, για περισσότερη δημοκρατία. Είναι και μια ευκαιρία για τους Ευρωπαίου συμπολίτε μα να μπορέσουν να ελέγξουν και πάλι τη ζωή τους, να ελέγξουν το τι τρώνε, το πώς μετακινούνται, πού κατοικούν, τι ενέργεια χρησιμοποιούν, ενώ οι κοινωνίε μας είναι τόσο κατακερματισμένες και διχασμένες σήμερα. Οπότε η υπόσχεση είναι βέβαια πάρα πολύ γερή, αλλά όσο πιο γερή είναι αυτή η υπόσχεση, τόσο πιο εύκολα μπορεί να προδοθεί. Η Πράσινη Συμφωνία δεν μπορεί να είναι ότι βάζουμε ένα άλλο όνομα και κάνουμε τα πράγματα όπως τα κάναμε μέχρι τώρα. Δεν μπορεί να είναι μόλις και μεταβίας λίγο παραπάνω, λίγο καλύτερα. Δεν μπορεί να είναι ο ίδιος προπολογισμό που τον αλλάζουμε λίγο δεξιά-αριστερά για να του δώσουμε διαφορετικό τίτλο χρειάζεται να κόψουμε με το παρελθόν. Σήμερα αυτό που χρειαζόμαστε είναι δημόσιες επενδύσεις 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ κάθε χρόνο σώσαμε τις τράπεζες, μπορούμε τώρα να σώσουμε και το κλίμα. Κυρίως εάν πρόκειται έτσι να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης και να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία. Εφόσον λοιπόν η Πράσινη Συμφωνία είναι να σώσουμε το κλίμα, να δώσουμε νέο δυναμισμό στην οικονομία μας, να δημιουργήσουμε απασχόληση, τότε η συμφωνία με το Μερκοσούρ δεν μπορεί να υπογραφεί από εμά. Η συμφωνία αυτή δεν έπρεπε καν να προβλέπεται, γιατί όλοι γνωρίζουμε και το έχουμε συζητήσει τι καταστροφή γίνεται στα δάση της Βραζιλίας δύο φορές σε σχέση με πέρυσι εξαιτία του Βασονάρο. Ξέρουμε επίσης σε τι βαθμό ο πρόεδρος αυτό σε καθημερινή βάση παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών, είτε παραβιάζει ελευθερίες των αγωνιστών, των αυτοχθόνων ή των ομοφιλόφιλων. Δεν μπορούμε εμείς ακριβώς το όνομα των αξιών της Ευρώπης, το όνομα του περιβάλλοντος και του κλίματος εμείς να υπογράψουμε μια τέτοια συμφωνία. Η συμφωνία αυτή, για να συνοψίσω, είναι ότι εξάγουμε γερμανικά αυτοκίνητα για να εισάγουμε ε, βοδινό κρέας και σόγια. Όχι, η Ευρώπη του Green Deal δεν μπορεί να είναι αυτό, γιατί μια τέτοια Ευρώπη είναι μια Ευρώπη η οποία συνεισφέρει στην παγκοσμιοποίηση του κακού φαγητού, της κακομεταχείριση των ζώων, της καταστροφής των δασών και της απορρίθμισης του κλίματος και η παγκοσμιοποίηση επίσης της εξαφάνισης των αγροτών στις χώρες Μερκοσούρ, όπως επίσης και στις χώρες της Ευρώπης. Ξέρουμε ποιο είναι το δικό μας αγροτικό μοντέλο, το οποίο εξαρτάται από φυτικές πρωτεΐνες που εισάγουμε. Ε, σε ένα αντίστοιχο της επικράτειας ολόκληρης της Γερμανίας. Οπότε πρέπει να σταματήσει η διαπραγμάτευση αυτή με τη Μερκοσούρ και πρέπει να ξαναδούμε την κοινή γεωργική μας πολιτική. Και η πρόταση που κάνετε, κύριε Χόγκαν, που είσαστε επίτροπο για τη Γεωργία, δεν μπορεί να αντιστοιχεί στην Πράσινη Συμφωνία, δηλαδή πιο εντατική Γεωργία, λιγότερου αγρότε, περισσότερα φυτοφάρμακα. Δεν μπορεί να είναι αυτή η κοινή γεωργική πολιτική τη Ευρώπη και του Green Deal. Να αλλάξουμε την ΚΑΠ, λοιπόν, να αλλάξουμε τι εμπορικέ συμφωνίε. Η Πράσινη Συμφωνία μπορεί να είναι μια καταπληκτική ευκαιρία για την Ευρώπη. Και η κυρία Φοντερ Λάιεν σήμερα το πρωί είπε ότι πρέπει να ακούμε του Ευρωπαίου πολίτε. Ε, του, λοιπόν. Δεν θέλουν τη συμφωνία αυτή με το Μερκοσούρ θέλουν να δρούμε υπεύθυνα με συγκεκριμένε δράσει υπέρ του κλίματο τη βιοπικιλότητα και τη δημοκρατία. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα θα δώσω το λόγο στο Συμβούλιο. Κυρία Υπουργέ, η κυρία αν έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, αυτή η προτινόμενη συζήτηση, η συζήτηση είναι πάρα πολύ ε, σημαντική. Έρχεται μια εβδομάδα μετά που παρουσίασε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Αναμφισβήτητα αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα περιβαλλοντικά και κλιματολογικά. Θα πρέπει να παίξει το ρόλο της η Ευρώπη ανταποκρινόμενη σε όλα αυτά. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, θα αμφισβητήσουν οι επόμενες γενιές γιατί δεν δράσαμε αποφασιστικά. Το status quo δεν αποτελεί επιλογή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ηγηθεί και να κινηθεί ομαδικά για να μεταμορφώσει τις κοινωνίες μας και τις οικονομίες μας, ούτως ώστε να ακολουθήσουν μονοπάτι πιο βιώσιμο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα περιγράψει τι έχει να προτείνει πλευρά πολιτική λεπτομερέστερα. Το Συμβούλιο δεν έχει το χρόνο, δεν έχει το χρόνο να συζητήσει και θα ήταν πρόημο για μένα να τοποθετηθώ τώρα σε αυτή τη φάση. Είναι πρώιμη φάση. Μπορώ μόνο να πω ότι το Συμβούλιο θα εξετάσει επικοδομητικά τι προτινόμενε πολιτικέ και τα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη τη Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Αυτή η στρατηγική σχετική αφορά κάθε πολι... τομέα πολιτική και θα απαιτήσει προσεκτική εξέταση και συντονισμό. Αυτό είναι το υπόβαθρο. Θα ήθελα τώρα να εστιάσω τα σχόλιά μου επί της εμπορικής συμφωνίας Μερκοσούρ. Είμαι βέβαιη ότι πολλά μέλη του Κοινοβουλίου έχουν ισχυρά συναισθήματα περί της εμπορικής συμφωνίας που συνήφθη με τη Μερκοσούρ. Ξέρω ότι συζητήσατε το θέμα πρόσφατα, Φερρυπίν μετά τις δασικές πυρκαγιές που κατέστρεψαν την περιοχή του Αμαζονίου. Πράγματι, αυτό είναι άκρως ανησυχητικό για όλους μας. Όπως εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η συζήτηση και στο Συμβούλιο για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ είναι ακόμα σε μια πρώιμη φάση. Είναι σαφές ότι επαρκής χρόνος θα απαιτηθεί για μια διεξοδική εξέταση τη συμφωνία που ήταν τα αντικείμενο τη διαπραγμάτευση. Ανησυχίε για την εμπορική συμφωνία με το Μερκοσούρ θα πρέπει να μπορούν να ευσταθούν ε, και σε σχέση με το θεματολόγιο μα για την Πράσινη Συμφωνία. Οι ανησυχίε είναι κατανοητέ. Μπορούν οι εμπορικέ συμφωνίε να συμβάλλουν στην επίτευξη στόχων. Δηλαδή να εξάγουμε τα πρότυπά μα και του στόχου βιωσιμότητα προ χώρε. Αυτό μπορούμε να πετύχουμε μπορούν να αποτελέσουν όχημα για να πιστούν οι άλλοι να εφαρμόσουν φιλόδοξου περιβαλλοντολογικού και κλιματολογικού στόχου και πολιτικέ και να αποτελέσουν ένα τμήμα μια παγκόσμια ανταπόκριση στην αλλαγή του κλίματο. Εκατομμύρια θέσει απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ζωή των ανθρώπων εξαρτάται από το εμπόριο. Πρέπει να εξασφαλίσουμε το ότι το εμπόριο μπορεί να λάβει χώρα, εξασφαλίζοντα ταυτόχρονα ότι υποστηρίζει βιώσιμη ανάπτυξη και του κλιματολογικού στόχου τη Ευρωπαϊκή Ενώσεως και συμβάλλει σε βιώσιμο μέλλον. Θα ήθελα να επενθυμίσω